αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμές Μάκερ, τον εισηγητή. Και θα καλέσω και τον κύριο Βέλα να κατέβει τον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η επένδυση στη φύση και τη βιοπικιλότητα θα πρέπει να είναι κομβική σε μια Ευρώπη ε, αϊφόρα χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη. Η βιοπικιλότητα είναι ανυπολόγιστη ε, και στα πλεονεκτήματα τα οικονομικά. Ένα από τα, τις έξι ε, θέσεις ε, εργασίας στην Ευρώπη εξαρτάται από τη φύση. Το Natura 2000 που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ε, μας ε, κοστίζει 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο εάν δεν λειτουργεί σωστά. Ε, είναι από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες απειλές η απώλεια της βιοποικιλότητας. Ωστόσο δεν τα πηγαίνουμε καλά στη στρατηγική μας. Σήμερα απέχουμε πολύ από τους στόχους του 2020. Παρά τα όσα γνωρίζουμε ε, ότι ε, αν κάνουμε τις σωστές προσπάθειες θα έχουμε επιτυχία και παρά το γεγονός ότι οι στόχοι είναι εφικτοί, η γενική εικόνα παραμένει πάρα πολύ ζωφερή. Μόλις 23% των ειδών και 16% των βιοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ε, εάν δεν γίνουν σημαντικές προσπάθειες θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σενάριο όπως το 2010 και δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε και το 2020 θα ξαναχάσουμε τη συμφωνία. Ποια είναι η κεντρική ιδέα της έκθεσής μου. Χρειάζεται επιγόντως περισσότερη πολιτική βούληση για να αλλάξει η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Καλύτερη εφαρμογή, ισχυρότερος έλεγχος και μεγαλύτερη ένταξη της βιοπικιλότητας σε άλλους τομείς της πολιτικής. Όλα αυτά είναι εκ των ουκάνευ. Επιπλέον, θα πρέπει όλοι οι ενεχόμενοι να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτό. Μέχρι και ο, ο πολίτης ως άτομος. Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους είναι σημαντικός κρίκος της αλυσίδας. Τώρα γίνεται ένας έλεγχος υγιές, ένα fitness check ε, των οδηγιών αυτών και εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι οδηγίες Το αντίθετο. Θα πρέπει να υλοποιούνται ή στο ακέραιο η αναθεώρηση θα σήμαινε ότι χαλαρώνουμε τη στρατηγική για τη βιοπικιλότητα και θα υπήρχε μια μεγάλη περίοδος ανασφάλειας ε, από πλευράς νομικής ασφάλειας εννοώ και αυτό θα αποδυνάμωνε την ευρωπαϊκή πολιτική για τη φύση. Επιπλέον, είμαι πεπισμένος ότι η αναθεώρηση σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση. Δεχομένω τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, αλλά κυρίως με την ελληπή υλοποίηση και εφαρμογή και έλεγχο τη οδηγίας ή των οδηγιών για τη φύση. Και δεν είμαι μόνος μου σε αυτή τη θέση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος υποστήριξε σχεδόν ομόφωνα την έκθεσή μου και πιστεύω ότι και όλο το Κοινοβούλιο αύριο θα στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, πάνω από 500.000 Ευρωπαίοι πολίτες αντιτάχθηκαν με την αθεώρηση των οδηγιών ε, μέσω μιας εξτατείας που λεγόταν Nature Alert Campaign και η οι Υπουργοί στις 16 Δεκεμβρίου τόνισαν ότι υποστηρίζουν ε, τις οδηγίες αυτές για τη φύση και ζητούν μια καλύτερη εφαρμογή και όχι αναθεώρησή τους, Υπουργοί Περιβάλλοντος. Και τέλος, ε, τα πρώτα ευρήματα του fitness check δείχνουν ότι οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά και τότε και μόνο τότε έχουν αποτέλεσμα και πιάνουν τόπο. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Κύριε Βέλα, την περασμένη Παρασκευή πήγαμε μαζί ε, επίσκεψη ε, στον οργανισμό λιμένος ε, της Αμβέρσας και είδαμε πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει εκεί την οικονομική ανάπτυξη με τη φύση. Χάρη σε ένα δίκτυο πράσινων διαδρόμων και πυρήνων ε, διαφυλάσσονται και τα συμφέροντα του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού στην Ευρώπη και παντρεύονται με την προστασία της ε, νίδας και της χλωρίδας στο λιμάνι και στον ποταμό Σχέλντε. Βλέπουμε λοιπόν από την πολιτική στην Αμβέρσα ότι αυτό που χρειάζεται δεν είναι αναθεώρηση των οδηγιών αλλά πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή των κειμένων. Και θα πρέπει να διευκολύνεται η υλοποίηση όλων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ιδιαίτερα με ε, καλύτερες και βελτιωμένες κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές και να φροντίσει αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να αναγνωρίζονται πλήρως και να γίνονται σεβαστές. Καλό την Επιτροπή να ακούσει όλα αυτά τα μηνύματα και κυρίως την ανασφάλεια που μπορεί να ε, προκληθεί από το fitness check. Δεν επιτρέπεται να χάσουμε και άλλο χρόνο. Αν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία το 2020 και να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να ποντάρουμε στην πλήρη εφαρμογή των οδηγιών. Κατά τα άλλα, περιμένω και προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμπληρωματικές δράσεις και νοτόμες λύσεις, έτσι ώστε να σταματήσει στην Ευρώπη η απώλεια της βιοπικιλότητας. Και χρειάζεται και διευρωπαϊκό δίκτυο πράσινων υποδομών, καθώς επίσης και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω απώλεια βιοπικιλότητας. Υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές και θα πρέπει να μην χάνεται η βιοποικιλότητα και να προστατεύεται η επικονίαση. Ε, διακυβεύεται η υγεία ίδια, η ευημερία ε, και η ζωή των μελλοντικών γενεών. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και οδησηγητές ε, θερμά για την ιδιαίτερη υποστήριξή τους και την επικοδομητική συνεργασία. Ήταν για μένα προνόμιο και τιμή η ευκαιρία που είχα να συνεργαστώ μαζί σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο κύριος Βέλ. Ο Επίτροπος ο κύριος Βέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή, τον συνάδελφο κύριο Ντεμεσμάκερ, για αυτήν την έκθεση που αφορά τη βιοπικιλότητα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που μπορώ να συνεισφέρω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι για το 2020 που αφορούν τη βιοπικιλότητα. Αύριο θα υλοποιηθεί αυτή η έκθεση και δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα προς τον έξω κόσμο όσον αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και για την ανθρώπινη ευμερία αλλά και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια ώρα στέλνει και ένα μήνυμα ανησυχίας. Πρέπει να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, το φυσικό κεφάλαιο και η έκθεση αυτή μπορεί να στηρίξει, να βοηθήσει και να επιταχύνει την πρόοδο έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι μας με ορίζοντα το 2020 για την βιοπικιλότητα. Το ερώτημα είναι γιατί μιλάμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν έχουμε φτάσει στην υλοποίηση των στόχων. Περιορίζεται η βιοπικιλότητα, συρρυκνώνεται και υπάρχει απώλεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την βιώσιμη οικονομικοκοινωνική μας ανάπτυξη αλλά και για την ευημερία. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και την επίπτωση των κλιματικών αλλαγών. Υιοθετήσαμε την ατζέντα πολύ πρόσφατα 2020 για την βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και θεωρούμε ότι η πολιτική πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε περίπτωση απαιτεί καλύτερη υλοποίηση. Πρέπει να κινητοποιήσουμε φορείς σε όλους τους τομείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας. Θα πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία το Natura 2000, τα δίκτυα, τα πράσινα δίκτυα, ιδιαίτερα για την προστασία των υδάτινων πόρων και για την χρηματοδότηση του Natura 2016. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει σήμερα πολύ σημαντικές απαντήσεις. Είδαμε τη συμμετοχή του κοινού. Πάνω από 500.000 ε, Ευρωπαίοι πολίτες έχουν κινητοποιηθεί. Και είδαμε ότι αυτή η πολιτική μας έχει σήμερα δώσει πολύ απτά αποτελέσματα. Το fitness check είναι σε κάθε περίπτωση μια ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερα οι οδηγίες που αφορούν τη φύση να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά τους στόχους για την βιοπικιλότητα. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την υλοποίηση, άλλα που αφορούν την τεχνογνωσία, τον καλύτερη εξάπλωση της εμπειρίας μας και βεβαίως κάποιοι τομείς χρειάζονται ειδική προσοχή. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι προετοιμάζουμε τις τελικές μας ε, προτάσεις οι οποίες είναι έτοιμες την Άνοιξη σε σχέση με το fitness check. Βεβαίως η οδηγία που αφορά τη φύση παίζει ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την απώλεια της βιοπικιλότητας. Δεν αρκεί όμως, πρέπει να γίνουν πολύ παραπάνω έτσι ώστε να προστατευτεί η βιοπικιλότητα και να υπάρξει ανάκτηση στους τομείς όπου υπάρχουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Πρέπει να πάμε πέρα από τα δίκτυα Natura. Να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα στην βιοπικιλότητα και βεβαίως να διευρύνουμε τους στόχους ε, της ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοπικιλότητας και να οδηγήσουμε σε μια πιο λογική και βιώσιμη ανάπτυξη και κατανάλωση. Οι στόχοι για την βιοπικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντικοί, όχι μόνο γιατί είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τη φύση και γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη. Πρέπει να τους ενσωματώσουμε στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό μας. Η ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση έχει εντοπίσει πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως τον αγροτικό, την δασοκομεία που αφορά το 80% των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο για την αλληλεία, την ανάπτυξη και το θέμα των εμπορικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, η απώλεια στο τομέα της βιοποικιλότητας πλήττει και άλλους τομείς και υπάρχουν και κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα καθώς και βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω το θέμα της ε, υιοθέτησης της οδηγίας για τα είδη τα οποία είναι χωροκατακτητικά. Και σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες σε αυτό το τομέα, καθότι αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες για την απώλεια βιοπικιλότητας. Προστασία συγκεκριμένων ειδών. Προετοιμάζουμε επιπλέον εργασία για την αναθεώρηση πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις για την προστασία της απώλειας βιοπικιλότητας διεθνώς, τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διεθνή απώλεια βιοπικιλότητας και πιστεύω ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε θετικά αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε με πιο μεγάλη αισοδοξία στους στόχους του 2030. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεμπάστα, έχετε ένα λεπτό εξ ονόμου της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έχουμε να κάνουμε με μία πλήρη έκθεση από πλευράς ανάπτυξης, τη Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο. Είχαμε προβάλει συγκεκριμένα αιτήματα οι στρατηγικές ανάπτυξης να μην υποστηρίξουν πολιτικές κατά της βιοπικιλότητας. Τίποτα να μην πλήξει την βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πιο ευάλωτες ε, κατηγορίες, δηλαδή τους ε, γεωργούς και αυτούς που ζουν στην Ήπεθρο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βιοπικιλότητα μειούμενη μπορεί να πλήξει όλα τα είδη, ακόμα και τον άνθρωπο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι η νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας. Αύριο θα υπερψηφίσουμε τη στιγμή που θα είναι η ναυαρχίδα μας η υπεράσπιση της ε, βιοπικιλότητας. Κύριε Σεβαστιά, πρέπει να καταλήξετε. Υπερβήκατε το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Λίντς, 1,5 λεπτό από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινά τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή και ειλικρινή συνεργασία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει ως ομάδα ε, μια ισχυρή αντίδραση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της βιοπικιλότητας. Και εδώ σας παραπέμπω και στο fitness check των δύο κεντρικών οδηγιών για την προστασία της φύσης. Ως συγητής από πλευράς του ΕΛΚ είμαι κατά α, ε, της αναθεώρησης οδηγίας. Και δεν επικρίνω τη νομική βάση αυτή καθ' αυτή. Αυτό που ζητώ είναι πολιτική βούληση και από τα 28 κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ε, είναι καλύτερη η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η έκθεση πρωτοβουλίας ε, θα πρέπει να εστιαστεί ε, στην ενδιάμεση αναθεώρηση με τη στενή έννοια και όχι να καλύψει όλη τη βιοπικιλότητα. Θέλω σαφή και συγκεκριμένη απάντηση από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό περιμένω. Ε, γι' αυτό αύριο ζήτησε κατά τμήματα ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για μια καλύτερη βιοπικιλότητα θα πρέπει φερόμενοι φορείς να ασχολούνται. Δεν θα πρέπει να αποφασίζεται ρήμη των ε, γεωργών και των αγροτών η βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Εγώ το θεωρώ λάθος. Τώρα μόλις αναθεωρήσαμε την κοινή γεωργική πολιτική δεν θα πρέπει να την καταδικάσουμε αμέσως. Αφήστε τα μέτρα τα καινούρια να ε, εφαρμοστούν, να δούμε τι χωλαίνει και αν χρειαστεί να γίνουν και προσαρμογές. Ε, θα ε, μπορούσε να υπάρχει μια δυνατότητα προστασίας της φύσης με συμβάσεις. Ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ προσπαθήστε να σέβετε το χρόνο σας γιατί έχουμε ήδη μεγάλη καθυστέρηση. Η κυρία Κάντενπαχ για δύο λεπτά εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, δύο μηνύματα. Πρώτον, θα πρέπει σοβαρά να προωθήσουμε τη βιοπικιλότητα και δεύτερον, Υπάρχει πολύ ε, σαφής δέσμευση του Κοινοβουλίου και θα το δείτε και αύριο στη ψηφοφορία που θα επιβεβαιωθεί ότι δεν χρειαζόμαστε αναθεώρηση των δύο οδηγιών για την προστασία της φύσης. Εμείς είμαστε πεπισμένοι, το δείχνουν και τα παραδείγματα καταφανώς, ότι εκεί που ε, σωστά εφαρμόζεται η νομοθεσία και σωστά υλοποιείται πιάνει τόπο. Η ε, αηφορία δηλαδή παράγεται στη βιοπικιλότητα και στη φύση. Τώρα, να ανοίξουμε όλα τα πακέτα και να φέρουμε τα πάνω κάτω δεν θα βοηθήσει, θα είναι αντιπαραγωγικό γιατί παράγει ανασφάλεια. Κύριε Επίτροπε, σας εκλυπαρούμε. Χρειαζόμαστε τη βιοπικιλότητα, το βίο, τη ζωή την ίδια αλλά αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι αναθεώρηση των οδηγιών. Τη δική σας υποστήριξη χρειαζόμαστε στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ στα κράτη-μέλη και στην παρακολούθηση και επιτήρηση, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα μεγάλο τμήμα των κρατών μελών σε πολλούς τομείς ε, δείχνει επιπολαιότητα και δεν εφαρμόζει σωστά τις οδηγίες. Βίωση σημαίνει ζωή. Ποικιλότητα είναι πολυμορφία. Κάθε μέρα χάνουμε 150 είδη. Καθημερινά στον κόσμο. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των εδαφών, με την ποιότητα των υδάτων, με την ποιότητα ε, των οικολογικών μας υπηρεσιών. Ας προσπαθήσουμε από κοινού στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουμε την ανάγκη της εφαρμογής αυτών των οδηγιών. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο λαός, οι πληθυσμοί το ξέρουν. Αυτά τα δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι πολίτες. Αυτή η βιοπικιλότητα θα πρέπει να αποκτήσει και βίο για πραγματική ζωή. Ούτε απλουστεύσει θέλουμε ούτε τίποτα. Αυτό μόνο ανασφάλεια θα φέρει για να μην πω επιδείνωση της κατάστασης. Μόνο από κοινού μπορούμε να εφαρμόσουμε τους στόχου μας μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μνίτσεσκα, μέρο τη ECR. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται. Η Πολωνία είναι μια πολύ πλούσια χώρα στον τομέα αυτό. Η έκθεση του κυρίου Μέκερ εστιάζει σε όλα τα προβλήματα αυτής της ε, στρατηγικής που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρ' όλα αυτά, η νομοθεσία για τα σχιστολιθικά αέρια πάει πολύ μακριά και αν υιοθετήσουμε αυτήν την νομοθεσία θα είναι αδύνατον να υπάρξει εξόριξη αυτού του αερίου. Η Πολωνία χρειάζεται ανεξαρτησία ενεργειακή, να μην εξαρτάται από την Ρωσία και θα πρέπει να στραφεί προς αυτήν την μέθοδο εξόριξης και το σχιστολιθικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι η ρογμάτωση είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται στις αρχές μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίνεκ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε μέτρα για να ανταποκριθούμε στους στόχους βιοπικιλότητας το 2020, όπως κάναμε το 2010. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο ε, εάν αλλάξουμε την νομοθεσία μας που είναι ο χρυσός κανόνας που προστατεύει τα, ιδιαίτερα τα πτηνά στο οικοσύστημά τους με βάση τη συναφή οδηγία. Χιλιάδες ήδη προστατεύονται και έτσι υπάρχουν οικονομικά ευεργετήματα. Μιλάμε για 300 δις ετησίως. Εάν αναθεωρήσουμε τις οδηγίες θα έχουμε νομική ανασφάλεια και θα αποκλίνουμε από τους στόχους βιοπικιλότητας. Χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Η προστασία βιοπικιλότητας έχει και οικονομικούς στόχους. Εάν χάσουμε τους στόχους μας, θα μας στοιχήσει 50 δις ετησίως. Αυτές τις υπηρεσίες θα χάσουμε. Και φυσικά θα πλήξουμε τη βιόσφαιρα και αυτό θα έχει επιπτώσει στην Ήπειρό μας. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε χρόνο, Επίτροπε. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ανταποκριθούμε στους στόχους του 2020. Θα συνεργαστείτε με το Συμβούλιο για την Προστασία της Βιοπικιλότητας. Ξέρουμε ότι επειδή δεν εφαρμόζουν την ομοθέσια τα κράτη-μέλη, γι' αυτό υπάρχει, εκεί υπάρχει και μεγάλη ρήξη και λυπούμεθα που το Συμβούλιο δεν είναι σήμερα εδώ να λάβει μέρος στη συζήτηση. Θα ε, τηρήσετε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να διώκονται και εκείνοι οι οποίοι δεν προστατεύουν την βιοπικιλότητα. Οι πολίτες προσβλέπουν σε εμάς οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι υπόλογες. Αυτά είναι βήματα που θα πρέπει να λάβετε για να προστατεύσετε τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Δεν θα δεχτώ μπλε κάρτα γιατί είμαστε πάρα πάρα πολύ καθυστερημένοι. Έχουμε ακόμα και τις ε, ουλίες ενός λεπτού. Η κυρία Μπόλιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ η βιοπικιλότητα περνάει κρίση στην Ευρώπη και αυτό το δέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει γίνει ακόμα σημαντική πρόοδος για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή τη συρρήκνωση της βιοπικιλότητας. Και βλέπουμε ότι ναι μεν υπάρχουν κάποια πρόοδος, η οποία όμως είναι ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση αυτή η αναθεώρηση της οδηγίας ε, για την φύση θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Οι κότοποι απειλούνται και πολύ λυπάμαι γιατί σε αυτήν την έκθεση δεν είναι σαφής η αντίθεση προς αυτήν την αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση. Το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία, δεν είναι τα κείμενα, αλλά η εφαρμογή τους, η υλοποίησή τους. Και ελπίζω αύριο να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στους 500.000 Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι πολύ δυνατά μας στέλνουν ένα μήνυμα όσον αφορά την προστασία και μας λένε «Ακούτε» και αυτό λέω και προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είχαμε εξαιρετικά καλή συνεργασία με τους σκιόδους. Αρωτιέμαι, τι κάνετε εδώ. Θα ακούσετε αυτούς όλους που μας λένε να μην αλλάξουμε κάτι. Φαίνεται ότι αυτά που ακούμε είναι σαφέστατα μηνύματα. Δηλαδή, έχετε εξαιρετικά θέματα, νομοθετείτε για πολύ σοβαρούς τομείς, αλλά δεν έχετε αποτελέσματα. Σταματήστε λοιπόν εδώ και ασχοληθείτε πολύ περισσότερο με την υλοποίηση, με τον έλεγχο. Ακούμε ότι υπάρχουν οπισθοχωρήσεις. Ξέρω ότι πιέζεστε αλλά εγώ θα ήθελα να πω και στον κύριο μας και όλοι εμείς εδώ μέλη του Κοινοβουλίου θέλουμε να σας στηρίξουμε. Θέλουμε να επιβιώσουμε, θέλουμε να προστατεύσουμε την φύση όλοι μαζί. Είναι ένας κοινό στόχος και εδώ θα αναφερθώ στην σύμβαση του όρχους. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούμε να μπορούμε να προσφύγουμε στα δικαστήρια να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εργαλεία έχουμε, ας τα χρησιμοποιήσουμε. Και εδώ από κοινού το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να δράσουν. Ο κύριος Αφρόντε. Η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική, εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε, εγώ ήμουν σκιώδης, υπάρχει σωρία προτάσεων εδώ. Θα την υποστηρίξουμε. Αύριο θα υπάρξει θετική έκβαση. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στους στόχους του 2020 για τη βιοπικιλότητα. Η μεσοπρόθεσμη έκθεση είναι καταστροφική. Δεν βρισκόμαστε ούτε καν κοντά στις στοχοθετήσεις μας βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν πολύ λίγα για να προστατεύσουν την βιοπικιλότητα, να προστατεύσουν τον πλούτο τους. Θα θέλαμε, Επίτροπε, να ε, τηρήσουμε την οδηγία περί ενδιαιτημάτων και πτηνών και να μην αλλάξουν οι οδηγίες αυτές. Η κυρία Γιούζο για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η προστασία της βιοπικιλότητας έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε εμάς. Γιατί ξέρετε ότι εμείς συνεισφέραμε στο Natura 2000 πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. Και αυτό αφορά και ε, το θαλάσσιο τομέα. Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό πλαίσιο και φτάσαμε σε στόχους. Δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα. Θα πρέπει να δεχτούμε την ενίσχυση και την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας που υπάρχει με βάση την πείρα μας. Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα ήταν ε, παλινοδρόμηση θα πρέπει να παραμείνει η νομοθεσία ως έχει. Το πιο σημαντικό θα ήταν η Επιτροπή με συνεργασία των κρατών μελών να προβάλλει σωστές κατευθυντήριες γραμμές, σαφής οδηγίας, που να μπορέσουν να ισχύσουν ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αντιφάσεις. Εμείς έχουμε μεγάλα προβλήματα ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, ύπαρξη λύκων που πλήττουν το ζωικό μας κεφάλαιο και αυτό έχει σημασία και στον τομέα των πτηνών όπου υφιστάμεθα μεγάλες απώλειες. Δυστυχώς ε, σταμάτησε, τελείωσε ο χρόνο μας. Μπριάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η βιοπικιλότητα επλήγει από τις κλιματικές αλλαγές, την μόλυνση του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Μιλάμε για μία ε, οικονομική αρχή που δημιουργεί θέσεις εργασίας μόνο στο ε, Natura 2000. Στην περίπτωση της ε, επικονίασης εκτιμάται ότι το κέρδος ε, ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ετησίως. Ε, ε ας σκεφτούμε τι συμβαίνει με τις πλημμύρες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εργασία μας όπου ε, προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια της δασοκομείας, της ε, γεωργίας και του κυνηγιού να βρούμε κοινέ λύσεις. Μας ενδιαφέρει και ο τομέας της αλληλείας καθώς και οι λιμένες και οι θαλάσσιοι, τα, οι χώροι που θα πρέπει να τύχουν προστασίας. Ο κύριος Γκερμπράντη. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Μετά την προηγούμενη στρατηγική που απέτυχε η ΚΤΡΑ, εγώ το 2011 ορίστηκα εισηγητής για τη βιοπικιλότητα και συμφωνήσαμε ότι τώρα θα άλλαζαν τα πράγματα. Εδώ μέσα σε αυτό το ημικύκλιο όλοι τονίζουμε την τεράστια σημασία που έχει η βιοπικιλότητα για την ανθρωπότητα. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά το πλήρες φάσμα. Και είπαμε ότι τώρα θα άλλαζαν τα πράγματα. Μεταρρυθμίσαμε τη ε, αλευτική πολιτική και πέτυχε ε, με μεγαλύτερη εφορία τι έγινε με την κοινή γεωργική πολιτική, με την πολιτική συνοχή. Εκεί αποτύχαμε και πάλι. Δεν έγινε πιο βιώσιμη. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα το 2016 στα μισά του δρόμου και ε, ένα συμπέρασμα ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει σοβαρά ε, στην επίτευξη της στρατηγική της για τη βιοπικιλότητα. Δεν ε, έχει νόημα να τα συνεχίζουμε ε, αυτά τα πράγματα έτσι με τον ίδιο τσαπατσούλικο τρόπο. Μην, Μην απογοητεύετε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους εσείς στο Συμβούλιο και η Κομισιόν και κάντε σημαντικά βήματα για τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ρίτ. Εμείς, το που ξέρουμε τη σημασία της προστασίας ε, του περιβάλλοντος και της άγριας φύσης στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα ωραία μονοπάτια της ε, χώρας μας και βεβαίως χρειάζεται νομοθεσία γι' αυτό. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να υπάρξει επιπλέον ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι καλύτεροι για να προστατεύσουν τους οικότοπους της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, είναι οι Βρετανοί πολίτες και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι με τις αλλαγές του κλίματος και επειδή ακριβώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τα άγρια είδη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καταστροφή των οικοτόπων, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε τους δρόμους και την άσφαλτο να καταστρέφει όλο και περισσότερες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ντεμές Μάκερ για την εργασία του. Αυτό το ανέφεραν και πολλοί άλλοι ομιλητές. Θεωρώ ότι η κατάρτιση αυτής της έκθεσης θα πρέπει να συνεισφέρει στην ε, ανάλυση της ε, κατάστασης στο περιβάλλον και για μελλοντικές αναθεωρήσεις. Δεν θα πρέπει να γίνει τώρα αναθεώρηση. Το κάθε πράγμα στο χρόνο του. Έχει σημασία να εφαρμόσουμε το πλαίσιο. Θα, δεν θα υπάρχει νομική ασφάλεια για την βιοπικιλότητα διαφορετικά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παγίδες που ελοχεύουν αν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει η Επιτροπή να ορίσει έναν διεξοδικό κατάλογο των χωροκατακτητικών αλόχθονων ειδών και να δούμε ποια είναι τα επικίνδυνα χωροκατακτητικά είδη όπως ορίζει η ΕΦΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα όπως ορίζει η έκθεση. Για τα χωροκατακτητικά είδη η κίνδυνη είναι όλο ένα και μεγαλύτερη, γι' αυτό θα πρέπει να αντικρούσουμε τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν πολλές απειλές στην ε, βιοπικιλότητα και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, προκλήσεις. Ο κύριος Χάιτεμα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τεράστια η πρόκληση για τον κόσμο να παράγει τρόφιμα, αλλά για να μειώσει και την πίεση στα ε, ε, και οικοσυστήματα. Ε, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι αγρότες και οι ανθοκόμοι σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ε, τροφίμων και με βελτίωση της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό πιστεύω ότι η μεγαλύτερη απειλή και ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η γεωργία και η ανθοκομία, αλλά η άγνοια και η μη Δεν υπάρχει μία λύση για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Με σύγχρονες μορφές γεωργίας βελτιώνουμε το ε, έδαφος και χρειαζόμαστε λιγότερη γη για παραγωγή ενός κιλού τροφίμων. Στην Ολλανδία γίνονται αυτές οι προσπάθειες στο Natura 2000 ε, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τη φύση. Μόνο με συνεργασία, με κοινή λογική, με ε, συμμετοχή των γεωργών και των αγροτών που ξέρουν τι τους γίνεται θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Κιώστινιέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απώλεια της βιοπικιλότητας δεν σημαίνει μόνο απώλεια φύσης, αλλά και απώλεια οικολογικού πλούτου. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο τα γνωρίζει αυτά τα θέματα και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη βιοπικιλότητα και για την οικολογία και για τη φύση. Η στρατηγική λοιπόν βιοπικιλότητας για το 2020 ε, δίνει σωστές οθήσει με τους έξι βασικούς τομείς και συμφωνούμε όλοι ότι εκεί που χωλαίνει το πράγμα είναι στην υλοποίηση. Δεν δείχνουν την ίδια προθυμία παντού στην Ευρώπη ε, να υλοποιήσουν όλοι αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό καλωσορίζω και την καλύτερη εφαρμογή της κείμενης οδηγίας. Τι να την κάνουμε την αναθεώρηση και χαίρομαι που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου το βλέπει έτσι. Δεν έχει να τη συζητάμε την αναθεώρηση. Ε, το βασικό πρόβλημα ποιο είναι και εδώ χρειάζεται να εστιάσουμε πολύ περισσότερο. Οι αγρότες δεν συμμετέχουν πάρα πολύ ε, σε ό,τι αφορά ε, το χαρακτηρισμό των ε, περιφερειών Natura 2000. Υπάρχει πρόβλημα με τις μονοκαλλιέργειες, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ευσυνείδητους αγρότες που το κάνουν με τρόπο πάρα πολύ φυσικό και είναι κρίμα να γίνονται όλα αυτά ερήμην τους και να τους ε, αναγκάζουμε ε, ε, να περιορίζουν το εισόδημά τους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν περισσότερο αυτοί οι αγρότες στη χάραξη πολιτικής, να τους ακούμε, να τους υποστηρίζουμε, γιατί και αυτοί στηρίζουν τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Ντόρφμαν. Για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή προβληματιζόμαστε εάν η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαφύλαξη ε, της βιοπικιλότητας είναι σκόπιμη και επαρκής. Θα πρέπει όμως να προβληματιστούμε και ε, στο εξής. Είναι εύστοχα αυτά που λέμε. Ε, υπάρχουν ορισμένα είδη πανίδα στην Ευρώπη που απαγορεύεται να θυρεύονται αλλά είναι μεγάλη απειλή Βλέπετε τι γίνεται με τις αρκούδες και με τους λύκους που αλωνίζουν στα βουνά μας γιατί λέει προστατεύονται. Ωραία. Ε, αυτή είναι η βιοπικιλότητα. Εγώ προέρχομαι από τις Άλπεις, κατάγομαι, από μια περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο οι λύκοι και οι αρκούδες που δεν αφήνουν σε χλωρό κλαρί τους αγρότες. Ε, και είναι πολύ δύσκολο να έχεις ζώα να βόσκουν ελεύθερα στο λιβάδι. Ε, στο μεταξύ έχουν επιτεθεί και σε ανθρώπους και καταλαβαίνετε ότι είναι τουριστική η περιφέρεια αυτή και δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Ε, έχουμε προγράμματα και ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην τοποθέτηση παγίδων για αυτά τα θυράματα, για αυτή την πανίδα καλή βιοπικιλότητα, αλλά θα πρέπει να συνάδει και με την ασφάλεια των πολιτών. Αλλιώς θα μας φάνε ο λύκος και η αρκούδα και αυτοί θα έρχονται όταν θα φεύγει ο αγρότης. Ο αγρότης φεύγει, ο λύκος και αρκούδα έρχονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτερλε, για ένα λεπτό. Θα σε ευχαριστώ. Βεβαίως η βιοπικιλότητα είναι κάτι που πρέπει να το προστατεύσουμε, είναι σημαντικό για το ανθρώπινο είδος και την δική μας επιβίωση. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε περισσότερη πολιτική βούληση για να δούμε γιατί η αποτελεσματικότητά μας είναι τόσο χαμηλή. Πεθαίνουν καθημερινά ήδη, εξαφανίζονται και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να το σταματήσουμε. Πλήττουμε το περιβάλλον, η γεωργία και άλλοι τομείς συνεχίζουν να καταστρέφουν το περιβάλλον. Πρέπει να αλλάξει ο προσανατολισμός. Η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να εστιάσει την βιώσιμη ανάπτυξη, την βιώσιμη γεωργία και την λογική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με το Catch the Eye. Κυρία Πέτμια, είναι η πρώτη. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε τις επιπτώσεις επί της οικονομίας μας για όλες αυτές τις αποφάσεις που αφορούν την Natura 2000. Είδαμε ότι πολλά είδη προστατεύτηκαν, είδη που βρισκόταν υπό εξαφάνιση. Και την ίδια ώρα 5.000 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιοπικιλότητα δεν απειλείται σε όλους τους τομείς. Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι το θέμα της απώλειας βιοποικιλότητας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ζουν κοντά στις προστατευόμενες περιοχές, λιγότερο από 20 χιλιόμετρα παραδείγματος χάρη από μια περιοχή Natura, είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Γι' αυτό και θα πρέπει να διευρύνουμε αυτά τα δίκτυα και τις πρωτατευμένες περιοχές. Στην Κροατία η ευαισθητοποίηση είναι μεγάλη και είναι εξάλλου και η χώρα που καλύπτεται από τεράστιες περιοχές Natura 2000. Ευχαριστώ πολύ δεν άκουσα το όνομά μου να εκφωνείτε. Σας ευχαριστώ πάντως που μου δίνετε το λόγο. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία νομοθεσία ε, η οποία κρίνεται επαρκής, αλλά έχουμε προβλήματα εκτέλεσης. Θα πρέπει λοιπόν να ρίξουμε το φταίξιμο στις κυβερνήσεις, γιατί για ένα λόγο ή άλλο, για κάποιο λόγο, στρέφουν τα νότα τους προς την νομοθεσία αυτή. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τη δράση αυτή κατά της φύσης, όπως ισχύει και για την παραβίαση ανθρώπων. Κύριε Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Γεωργία διαδραματίζει αναμφισβήτητα ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας. παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των αγροτών της ευρώπης. δεν μπορεί ο αγροτικός πληθυσμός των περισσότερων χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης να απολαμβάνει ελάχιστους ή και μηδενικούς φόρους στο αγροτικό πετρέλαιο και την ενέργεια ενώ την ίδια στιγμή στην ελλάδα η τρόικα και τα μνημόνια να επιβάλλουν δυσβάστακτη αύξηση φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο καθιστώντας την αγροτική παραγωγή όλο ένα και λιγότερο ανταγωνιστική την ώρα λοιπόν που οι έλληνες αγρότες παλεύουν να σώσουν το ασφαλιστικό και τον ογά δέχονται ακόμη μια πισόπλατη μακεριά καθώς κύριε βέλλα μετά από απόφαση της κομισιόν και της επιτροπής διεθνούς εμπορίου της ευρωβουλής δρομολογείται η ελεύθερη και αδασμολόγητη εισαγωγή στην ελλάδα 70.000 τόνων λαδιού από την τινησία για την επόμενη διετία και μάλιστα αναδρομικά από 1 η 1 2016 στεκόμαστε λοιπόν δίπλα στους χυμαζόμενους από το μνημόνιο αγρότες μας και θα δώσουμε τη μάχη ώστε να σταματήσει η φτωχοποίηση των ελλήνων αγροτών. Η κυρία Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι δεν αμφισβητεί κανείς ότι η βιοπικιλότητα είναι πολύτιμο αγαθό, άξιο προστασίας και βεβαίως θα πρέπει να διαφυλάσσεται. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Υπάρχουν απαιτήσει που θα πρέπει να είναι ισορροπημένες σε σχέση με άλλους στόχους. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η ε, γεωργία και η δασοκομεία που παίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαφύλιξη της βιοπικιλότητας. Από επιστημονική άποψη ενδιάμεση έκθεση δεν επιτρέπει ε, ουσιαστική ε, αξιολόγηση της κατάστασης. Δεν είναι σοβαρό αυτό που λέει ότι 80% των δασών δεν είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία από τα 28 κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε χρειάζεται σαφής ε, ε, ε βελτίωση και στην επικοινωνία και στη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των γεών και ε, συλλογή πραγματικών στοιχείων. Ο κύριος Φεραίρα. Ευχαριστώ κατακαιρμάτιση των οικοσυστημάτων καθώς και των φυσικών ε, χώρων. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη όλα αυτά ορίζουν και υποσκάπτουν τη βιοπικιλότητα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Δεν χρειάζεται μία ενίσχυση των μέσων για να ε, ανασχέσουμε τη μείωση της βιοπικιλότητας, αλλά χρειάζεται και ενίσχυση της, ε, του αγροτικού κόσμου, έτσι ώστε να μην υπάρχει ερήμωση των χωριών, να καταπολεμήσουμε τα χωροκατακτητικά είδη και να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα την Ατούρα 2000. Επίσης χρειάζεται ενίσχυση του προγράμματος Life και Life Plus. Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα που προβάλαμε μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Βεβαίως, στηρίζω να προστατεύσουμε την πλούσια βιοπικιλότητα της περιοχής μου. Και βεβαίως έχουμε δικούς υδάτινους πόρους και υδρότοπους στην περιοχή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν και στηρίζω και συμφωνώ με την περισσότερη τις περισσότερες από τις προτάσεις αυτής της έκθεσης. Όπως όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα. Χρειάζεται όμως και κοινή λογική και η έκθεση αυτή προτείνει γραφειοκρατία. Ενώ χρειαζόμαστε περισσότερους αληθικούς πόρους, βλέπουμε ότι εδώ προτείνει περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική. Προτείνει περισσότερη συγκέντρωση και όχι τοπικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Κατσιάη και στραφόμαστε και πάλι σε εσά κύριε Επίτροπε, κύριε Βέλα. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη μεγάλη του δέσμευση και υποστήριξη της βιοπικιλότητας και της φύσης. Θεωρώ ότι όταν εγκριθεί το ψήφισμα μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Δεκέμβριο θα βοηθήσει στο να φτάσουμε στη, στους στόχους της βιοπικιλότητας. Και η ενδιάμεση αναθεώρηση ε, δείχνει ότι χρειάζεται ολοκλήρωση των στόχων της βιοπικιλότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε στους στόχους της βιοπικιλότητας. Λαμβάνω υπόψη και τον ε, όγκο της βιοπικιλότητας και εντάσσοντας τους στόχους σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και μετατρέποντας αυτό το ψήφισμα σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικών και χρηματοδότησης. Χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομοθεσία και αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Συμφωνώ και με πολλούς ομιλητές που εξέφρασαν την άποψη ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, για την εφαρμογή. Όπως είπε και ένα μέλος, θα πρέπει να ε, επιταχυνθεί η εφαρμογή. Η κυρία Μπόιλε με ρώτησε κατά πόσο μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια συλλογική ευθύνη και απόφαση με βάση το fitness check το οποίο θα ολοκληρωθεί. Θα κοιτάξουμε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για την επίτευξη των στόχων 2020 έλαβα υπόψη αυτά που είπε η κυρία Όκιν, δέχομαι αυτά που προείπατε, αλλά νομίζω ότι όλοι οι επίτροποι και ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς έχουν ταχθεί υπέρ της φύσης και της βιοπικιλότητας. Πολλά μέλη είπαν ότι θα πρέπει οι αγορότες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο επίτευξης των στόχων της βιοπικιλότητας. Το έχουμε τονίσει αυτό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενδιάμεση έκθεση που δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι καθυστέρησης. Δεν μιλάμε μόνο για την εφαρμογή Μία από τις αιτίες δεν έγκυται στη γεωργία, αλλά στις κακές πρακτικές στη γεωργία με βάση την ΚΑΠ όπως έχει οριστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε μέσα βιοπικιλότητα σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να ορίσουμε και, το πώς θα ε, εκμεταλλεύονται τα αγροκτήματα και η αγροτική γη γενικότερα. Θα επιτευχθούν οι στόχοι της βιοπικιλότητας και στον αγροτικό τομέα κατά αυτόν τον τρόπο. Και όπως είπε και ο κύριος Κόστιγκερ, η κυρία Κόστιγκερ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγροτικό τομέα. Και θα ήθελα να πω ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες, αλλά είμαστε και αισιόδοξοι γιατί είναι ανεπαρκής η πρόοδος, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι έχει επιτευχθεί. Έχουμε ορίσει ένα πλαίσιο εργασίας, έχουμε θετική πείρα και εμπειρίες και μπορούμε να υποστηρίξουμε τις αποφάσεις μας. Επίσης έχουμε ένα διευρυνόμενο δίκτυο πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων. Θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό για να φτάσουμε στους ε, στόχους. Οι οδηγίες ε, στις οποίες προαναφερθήκατε δεν είναι αυτός σκοπός είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στους στόχους του 2020. Και αυτό μπορεί να γίνει και με την ενδιάμεση έκθεση μέσα σε μια γενικότερη συνεργασία για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ.